ρύθμιση σύμφωνα με το άρθρο 74 το περιεχόμενο θα περιλαμβάνεται στα πρακτικά της συνεδριάσεως αυτής και θα το ελέγξετε. Πήρα επίσης πληροφορίες από την ομάδα των πασίνων, την Ευρωπαϊκή Ελεύθερη Συμμαχία, ότι ο κύριος Φίλιπ Λάμπερτς αντικαθιστά την Εύα Ζολή στην Οικονομική Επιτροπή. Θέλετε να κάνετε μια παρατήρηση πάνω στην ανακοίνωση της ομάδας των Πρασίνων. Όχι. Αλλαγές τώρα στην ημερήσια διάταξη. Κυρίες και κύριοι, θα ξεκινήσω από τη Δευτέρα η ομάδα των φιλελευθέρων, όχι διορθώνω, η ομάδα των σοσιαλιστών και δημοκρατών ζήτησε η έκθεση Γκάλο να μην τεθεί προς Αφορά την πνευματική ιδιοκτησία. Ο κύριος Σούλτσο θέτει το ερώτημα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Πρόεδρε, η κοινοβουλευτική μα ομάδα ήδη στην διάσκεψη των Προέδρων την προηγούμενη εβδομάδα επεσήμανε ότι η έκθεση Γκαλό είναι πολύ επίμαχη έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας στο Σώμα, στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Όσον αφορά την περαιτέρω εξέταση αυτής τη έκθεσης, θα έπρεπε για άλλη μία φορά να εξεταθεί σε βάθο. Έχουμε μπροστά μα το εξή. Αυτή η έκθεση, σύμφωνα με τις νέες διεργασίες βάσει του κανονισμού μας, θα πρέπει να εισαχθεί, να ψηφιστεί, αλλά έχουμε ήδη άλλες εναλλακτικές ε, άλλα εναλλακτικά ψηφίσματα τα οποία τίθενται σε ψηφοφορία. Και εξάλλου από την κατάσταση όπως διαμορφώνεται είναι πολύ επίμαχο να προβλέψει κανείς. Εγώ τολμώ να πω ότι κανένα ψήφισμα δεν θα τύχει πλειοψηφία στο τέλος τέλος. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το άλλο θέμα είναι ότι εντωμεταξύ μάθαμε ότι στον τομέα των δικαιωμάτων, των πνευματικών δικαιωμάτων, οι πρωτοβουλίε της Ευρωπαϊκής Επιτροπής θα υποβληθούν τις επόμενες ημέρες. Άμεσα δηλαδή στο προσεχές μέλλον. Και έτσι νομικά έχει ληφθεί η απόφαση οδηγίες ε, νομικά να προωθηθούν. Δηλαδή αυτό τι σημαίνει. Εμεί, σε μια χρονική στιγμή όπου θα νομοθετούμε, θα νομοθετήσουμε, θα ψηφίσουμε για μια έκθεση ιδίας πρωτοβουλίας που σίγουρα θα θεωρείται μετά ανεδαφική και ξεπερασμένη από το νομοθετικό έργο που θα ακολουθήσει. Γι' αυτό ζητούμε να αποσυρθεί από την ημερησία διατάξη έκθεση. Σας ευχαριστούμε πολύ κύριε Σούλτς. Υπάρχει κάποιος που θα ήθελε να λάβει τον λόγο τώρα υπέρ αυτού του αιτήματος. Eh. Ναι, υπέρ, παρακαλώ, έχετε τον λόγο. Ε. Ευχαριστώ, Δεν μπορούμε να αποδεχθούμε ένα νέο αίτημα αναβολής της ψηφοφορία επί της εκθέσεως της Γκάλο. Είναι λάθος να λέμε επί της ουσίας ότι δεν υπάρχει απαιτούμενη συνένεση. Η έκθεση αυτή είναι αποτέλεσμα πολλών συμβιβασμών που έγιναν αντικείμενο συζήτησης για πολλούς μήνες επί του τύπου. Να μου επιτρέψετε να σας υπενθυμίσω ότι ψηφίστηκε στην Επιτροπή Νομικών Υποθέσεων στις αρχές του μηνός Ιουνίου. Έγιναν περαιτέρω συζητήσει μετά από τις τρεις αναβολές οι οποίες δόθησαν και αυτή τη φορά δεν υπάρχει πραγματικά καμία αιτία, κανένας λόγος αναβολής εκτός μόνο για να επιτρέψουμε σε ορισμένες πολιτικές ομάδες να βρούνε μια εσωτερική, αν θέλετε, μορφή συνένεσης. Δεν είναι αυτό όμως το γενικό συμφέρον. Το γενικό συμφέρον καλεί να ψηφίσουμε την έκθεση αυτή πρωτοβουλία, η οποία σε καμία περίπτωση δεν βρίσκεται σε αντίθεση με τις μελλοντικές νομοθετικές ρυθμίσεις. Η έκθεση αυτή απλά καλή την εφαρμογή των ε, υπαρχουσών νομικών ρυθμίσεων και πέραν τούτου τίποτα. Ευχαριστώ. Λοιπόν, είναι μια άποψη η οποία ήταν υπέρ του να διατηρηθεί η έκθεση αυτή στην ημερήσια διάταξη. Εγώ δεν έθεσα αυτό το ερώτημα όμως. Εγώ σας ζήτησα ποιος θέλει να υποστηρίξει τον κύριο Σούλτς και την πρότασή του. Κύριε Σπερώνη, όχι, ο κύριος Κομπεντήτ. Κυρία Γκάλο, έχω την αίσθηση ότι ο συνάδελφος Σούλτς είπε τα σωστά πράγματα, δηλαδή δεν υπάρχει πλειοψηφία και θα καταψηφίσει την έκθεσή σας και η ομάδα των φιλελευθέρων. Ας μην λοιπόν αποδείξουμε για μια ακόμη φορά ότι δεν υπάρχει απαιτούμενη πλειοψηφία. Υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω συζήτηση ε, σε όλες σχεδόν τις ε, πολιτικές ομάδες, εκτός από την δική σας, πολύ αμφιβάλλω βέβαια. Πάντως το θέμα αυτό στις περισσότερες πολιτικές ομάδες είναι πάντα υποσυζήτηση και δεν υπάρχει ξεκάθαρη πλειοψηφία. Για μία ακόμη φορά λοιπόν ο κύριος Σούλτς ζητά κάτι το ιδιαιτέρως λογικό. Για μία ακόμη φορά. Ζητώντας την αναβολή αυτής της νομοθετικής πρωτοβουλία. Σα ευχαριστώ και ολοκληρώνουμε έτσι τις διαδικασίες ε, με τα επιχειρήματα υπέρ και κατά. Και τώρα θα ψηφίσουμε. Ψηφίζουμε λοιπόν αίτημα της Σοσιαλιστικής Ομάδας. Με άλλα λόγια, το αίτημα του κυρίου Σούλτς. Όσοι είναι υπέρ του αιτήματο των Σοσιαλιστών. Ευχαριστώ. Κατά. Η πλειοψηφία είναι κατά του αιτήματο που διατυπώθηκε από τον κύριο Σούλτς Αλλά εντάξει, θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Θα ελέγξουμε ηλεκτρονικά. Άρχεται η ψηφοφορία ηλεκτρονικά. Παρακαλώ. Wszyscy głosowali. Ψηφίσατε όλοι και όλες. Ένας ψηφοφορίας. Και έτσι δεν εγκρίθηκε το αίτημα. Η πλειοψηφία ήταν εναντίον. Καταψηφίστηκε το αίτημα. Και παραμένει λοιπόν το θέμα εγγεγραμμένο στην ημερήσια διάταξη προς συζήτηση. Περνάμε τώρα στην Πέμπτη. Και μια και επειδή δεν υπάρχουν αλλαγές, σε σχέση με την ε, Τρίτη και την Τετάρτη. Την Πέμπτη τώρα οι συντηρητικοί και μεταρρυθμιστές ζήτησαν σε σχέση με την πρόταση ψηφίσματος όσον αφορά τις, ε, την ε, λήψη στην προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στην δημοκρατία του Κονγκό. Εδώ γίνεται λόγος για την αναβολή ακριβώς της ψηφοφορίας δηλαδή της πρότασης ψηφίσματος και είναι μια πρόταση της ομάδας ECR. Ο κύριος Μπράτμπορν έχει τον λόγο, παρακαλώ. Έχετε τον λόγο, παρακαλώ. Ευχαριστώ, πρόεδρο. Εξ ονόματος της πολιτικής μου ομάδας θα ήθελα να ζητήσω την αναβολή της ψηφοφορίας την Πέμπτη. Και αναφερόμεθα όχι στα υπόλοιπα θέματα, αλλά μόνο στην ψηφοφορία. Εσείς στην αρχή αυτής της συνεδρίασης είπατε τα πιθανά προβλήματα τα οποία θα αντιμετωπίσουν τα μέλη την Πέμπτη για να μπορέσουν να επιστρέψουν στις χώρες τους. Και γνωρίζω πολλά μέλη που θα φύγουν την Τετάρτη από εδώ για να μην δημιουργηθεί πρόβλημα. Συνεπώς είναι πολύ λογικό να ζητήσουμε μια αναβολή μόνο δύο εβδομάδων και να ψηφίσουμε στην μήνυ Ολομέλεια στι Βεξέλλε. Ευχαριστώ πολύ. Ποιοι είναι υπέρ της προτάσεως του κυρίου Μπράντμπορν. Ποιοι είναι υπέρ. Είναι ασυνήθιστη αυτή η συνεργασία, αλλά παρόλα αυτά η δική μου κοινοβουλευτική ομάδα ήδη την προηγούμενη εβδομάδα είχε προτείνει την Πέμπτη να μην γίνουν ψηφοφορίες. Και αυτό επειδή δεν έχουμε υπέρ, όπως φοβόταν ο κύριος Ντόρ, το δικαίωμα των Γάλλων εργαζομένων σε απεργία να τον αμφισβητήσουμε. Θα θέλαμε όμως να διασφαλίσουμε ότι δεν θα έχουμε τόσους πολλούς εργαζομένους από την Γαλλία ή την Γερμανία που θα καταβάλουν προσπάθειες ώστε η μεταφορά, ιδιαίτερα δαπανηρή μεταφορά των Ευρωβουλευτών και των συνεργατών τους να μπορέσει να λειτουργήσει και έτσι να υπονομευθεί εντός εισαγωγικών η απεργία. Από ό,τι γνωρίζω, από ό,τι πιστεύω στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, σίγουρα υπάρχει υποστήριξη για αυτή την λογική προσέγγιση, θα έλεγα. Και η δική μου κοινοβουλευτική ομάδα είναι υπέρ τη αναβολή αυτή τη ψηφοφορία. Ευχαριστώ. Πρόεδρο, σα ευχαριστώ πολύ. Τώρα κάποιο που θα λάβει τον λόγο εναντίον, ο κύριο Σπερώνη, κατά του αιτήματο. Το θέμα δεν είναι να ψηφίσουμε για μια νομοθετική πρόταση. Έχει λοιπόν μια σημασία θα έλεγα διαφορετική. Αυτή η απεργία τώρα θεωρώ ότι θα θίξει εν πολλής όλες τις πολιτικές δυνάμεις προφανώς που είναι παρούσες σε αυτό το κοινοβούλιο. Δεν είναι κάτι που θα θίξει μόνο τους αριστερούς ή μόνο τους δεξιούς. Μία θα έλεγα μειωμένη αντιπροσωπευτικότητα λοιπόν είναι κάτι το οποίο μας διασφαλίζει τη δυνατότητα ψηφοφορίας. Ποιοι είναι υπέρ λοιπόν της προτάσεως. Ποιοι είναι κατά του αιτήματο του κυρίου Μπραντφορντ. Ηλεκτρονικός έλεγχος. Ξεκινάει η ψηφοφορία. Ψηφίσατε όλοι. Τέλος. Λοιπόν, η πλειοψηφία είναι υπέρ της προτάσεως του κυρίου Μπράτμπορν, της αναβολής της ψηφοφορίας την Πέμπτη. Συνεπώς δεν θα υπάρξει ψηφοφορία για τη συγκεκριμένη έκθεση την Πέμπτη. Λοιπόν, περνάμε τώρα στη σημερινή ημερήσια διάταξη. Προβλέπεται η συζήτηση για την έκθεση της κυρίας Κριστίν Τεβεράκ σχετικά με την πρόληψη και την διερεύνηση των αεροπορικών ατυχημάτων. Έχετε το λόγο κύριε Ντεβεράκ. Πρόεδρε, κύριε Πρόεδρε, Πρόεδρε, δεν κατάλαβα τι έγινε με την ψηφοφορία. Ψηφίσαμε για την ημερήσια διάταξη που αποφασίστηκε στη διάσκεψη των Προέδρων ή κατά. Κατά. Ε, Οπότε δεν θα συνεδριάσουμε την Πέμπτη.